Βαϊ- ε, Witam Κυρίες και κύριοι, λέει ο Πρόεδρος, προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Καθίστε. Όλοι βιαζόμαστε για να προλάβουμε τρένα, αεροπλάνα, να φύγουμε τα αυτοκίνητά μας. Ε, αυτό να μην το ξεχνάμε. Η πρώτη ψηφοφορία τώρα. Μαλάουι και λοιπές αφρικανικές χώρες. Έχουμε ένα κοινό σχέδιο ψηφίσματος. Μετά είναι παραγραφό 3 με την τροπολογία 3 υπέρ. Κατά.